σύμφωνα με το άρθρο 74 ε, του κανονισμού μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω ε, τα κείμενα που εγκρίθηκαν, δέκα τον αριθμό ε, και στα σημερινά πρακτικά θα δημοσιευθούν οι επικεφαλίδες. Ερχόμαστε τώρα στην έγκριση της σημερινής διάταξης ή στην τροποποίησή της και στη διάταξη των εργασιών.